Ε, έχουν αυξηθεί ε, στο 26%. Όσον αφορά την περιφερειακή κάλυψη, εδώ υπάρχουν ε, κάποιες ελλείψεις. Ωστόσο, εξετάζουμε τις δραστηριότητά μας και την περιφερειακή του εμβέλεια. Για παράδειγμα, το ΕΦΣΙ δείχνει ότι η γεωγραφική διαφοροποίηση βελτιώνεται. Η Ιταλία, η Γερμανία και η Γαλλία έπεσαν τα ποσοστά. Ε, ωστόσο, αν τα συγκρίνουμε με το μερίδιο του ΑΕΠ, η αριθμοί είναι πολύ διαφορετική. Για παράδειγμα, η Ελλάδα, η Εστονία, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία και η Λιθουανία είναι οι βασικοί ε, παραλήπτες το 2018, εάν κάνουμε ακριβώς αυτή τη σύγκριση με το ΑΕΠ. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας καταλήξω λέγοντας ότι η ΕΤΕΠ εξεπλήρωσε τους στόχους της. Ε, το, μέσω του σχεδίου Juncker μπορέσαμε να συμβάλλουμε σημαντικά στην αύξηση της απασχόλησης και την ανάπτυξη οικονομίας στην Ευρώπη. Είμαστε η Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι υπερβαίνουμε τα εθνικά συμφέροντα ε, και είμαστε ένα υπόδειγμα της ε, Ευρώπης εν δράση θα συνεχίσουμε να κινητοποιούμε, να απελευθερώνουμε συγγνώμη, επενδύσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη ε, ασχολούμενοι με την ανάπτυξη των υποδομών σε όλη την Ευρώπη και αναβαθμίζοντας το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, παγκοσμίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χόιερ. Ο Επίτροπος Κατάινεν έχει το λόγο, παρακαλώ. Καταρχάς, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώργ Πυρίνσκι, τον εισηγητή και άλλους ευρωβουλευτές που συμμετείχαν στις εργασίες για την εκπόνηση της έκθεσης αυτής. Ε, είναι εξαιρετική η έκθεση αυτή. Όλοι γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι απαραίτητο εταίρος για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, καινοτομίε σε διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης, δράση για το μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, και άλλες επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την φιλόδοξη στρατηγική για την κλιματική δράση που ανταποκρίνεται στην προσήλωση των θεσμικών οργάνων. Επίσης, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή αποδοτικότητα, ε, ε, ο εστιασμός σε προϊόντα υψηλής ποιότητας ε, είναι στοιχεία κλειδιά όπως είναι και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νέους τομείς, όπως είναι ε, η τεχνητή νοημοσύνη ή η κυκλική οικονομία. Είναι απαραίτητο να έχουμε σωστή αντιστοίχηση ανάμεσα στις ε, χρηματοδοτικές ανάγκες και στα διαθέσιμα μέσα. Αυτό λοιπόν είναι μια συνεχιζόμενη πρόκληση για την τράπεζα, διότι η οικονομία γύρω μας αλλάζει. Στο πλαίσιο του Brexit ε, επικροτούμε τις προσπάθειες ε, της τράπεζας ε, να διασφαλίσει να μην επηρεαστούν οι δανειοδοτικές της ενέργειες. Ε, συνεργαζόμαστε στενά εντός της Επιτροπής για να βρούμε μια καλή λύση για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μετά το 2020. Εννοείται ότι η ΕΤΕΠ θα συνεχίσει να προωθεί τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και μετά το 2030. Σας ευχαριστώ. Σας ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Το λόγο έχει ο κύριος Στάρτμουθ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να αλλάξω τα λόγια του περίφημου λόγου του Μάρκου Αντωνίου από τον ε, ο Σέξπιρ, έρχομαι να φτιάξω την τράπεζα και όχι να τη θάψω. Ε, κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει καλύτερο ισοζύγιο, ισχυρότερο ισοζύγιο από ότι η Deutsche Bank ε, αυτή τη στιγμή. Η Βρετανική κυβέρνηση έχει 16% μετοχές με αξία 39 δις ευρώ. με αυτή την αξία να παραμείνει. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ή να προσκοληθούμε σε στερεές εμπορικές αρχές. Αυτό να μην ε, λόγω πολιτικών ε, επιταγών. Τα αιτήματα για την πολιτικοποίηση του δανεισμού θα πρέπει να να, να, μην τα υπακούσουμε και να αντισταθούμε σε αυτά, ιδιαίτερα εφόσον αυτά προέρχονται από, τους, ε, από τα πράσινα κόμματα και όσους εκεί συχνάζουν. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι εξ ονόματος του ΕΛΚΑ, ο κύριος Ντόιτς. Κύριε Πρόεδρε, σας, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν θέλω να είμαι εξαιρετικά ευγενικό, αλλά θέλω να, πραγματικά να συγχαρώ τον κύριο Πυρίνσκι για την σπάνια ποιότητα έκθεση, έκθεση του. η οποία συνοψίζει τα όσα έχει συμπεράνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια ε, σε σχέση με την ΕΤΕΠ και επίσης σέβεται και αντικατοπτρίζει τις επικρίσεις που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Υπάρχουν κάποια προβλήματα και υπάρχουν κάποια πράγματα που λείπουν, όπως λέει η έκθεση, αλλά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λειτουργεί ορθά, λειτουργεί όπως οφείλει. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι βασικά μια τράπεζα. Υπάρχουν προβλήματα δανεισμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση οι χώρες μάλλον που ήταν μέλη πριν το 2004 είναι σχεδόν αποκλειστική ε, δικαιούχη της δανειοδοτικής πολιτικής της και γι' αυτό θεωρούμε πως είναι απαραίτητο να επεκταθεί ο δανεισμός στις ε, υπόλοιπες χώρες μέλη και στα Δυτικά Βαλκάνια. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ε, καλωσορίζω τον κύριο Τακατάιναν και τον κύριο Χόγε. Σας ευχαριστούμε που είστε παρόντες σε αυτή τη συζήτηση και να ευχαριστήσω και να συγχαρώ και τον συνάδελφο Πυρίνσκι διότι σε αυτή την έκθεση έβαλε όλη, όλες τις γνώσεις και είχε εμβαθύνει στα περίπλοκες δραστηριότητες της ΕΤΕΠ, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη ότι Ε, και το ελεγκτικό συνέδριο μπορεί να ε, επιβλέψει αυτές τις διαδικασίες. Impact εδαφικός αντίκτυπος. Είπατε το 2018 θα σημαίνει σημαντική πρόοδο. Και ήδη βλέπουμε κάποια σειρά χωρών που είδαμε πως εδώ ήταν αυτές οι χώρες πέμπτες, πέμπτες δεν ξέρω αν η τέταρτη είναι η Ισπανία, η Ιταλία. Είναι όλες οι χώρες μαζί. Ε, τότε θα ε, είναι ε, εντάξει. Ε, δεύτερον, μεταναστευτικό φαινόμενο. Και πάλι έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Όπως είπαμε για την Αφρική, για να μην μιλήσουμε για τη Μέση Ανατολή, έχουμε προβλήματα γιατί τα μικροδάνεια για τις μικροεπιχειρήσεις ε, έχουν προβλήματα. Ε, η τράπεζά σας έχει ε, συνάψει διάφορες συμβάσεις, όμως όταν τα δούμε λεπτομερώς θα δούμε ότι τα περισσότερα είναι μηδενικά. Γιατί, και αυτό μας ανησυχεί, γιατί δεν πρέπει να επιτρέψουμε η ΕΤΕΠ να είναι τράπεζα για τις πολιτικές, τις αναπτυξιακές των βασικών μας συνομιλητών. Δεύτερον, Οι startup ζητάνε χρηματοδότηση. Ε, και τέλος, είχα την έκπληξη ότι δεν μετρώνται οι θέσει απασχόληση που δημιουργούνται από αυτά τα project. Δεν υπάρχει κανένα τρόπο να δούμε ποιο είναι ο αντίκτυπο στην απασχόληση αυτών των project. Νομίζω πω θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα να αρχίσει να μετρά και τι θέσει απασχόληση που δημιουργεί. Παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο μιλίας. Επόμενος ομιλητής εκ μέρους του ECR, ο κύριος Τσαρνέσκη, για ένα λεπτό. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Καταρχήν θα πρέπει να πει ε, ότι η τράπεζά σας δεν είναι policy maker αλλά policy taker. Δηλαδή όλα τα θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή τελικά χρηματοδούνται από τους ιδίους πόρους των χωρών μελών. Και η ΕΤΕΠ τελικά θέτει τις δικές της πολιτικές, ε, τους τις της πολιτικούς ε, στόχους το σχέδιο Juncker ε, και το ΕΦΣΑ. Εδώ υπάρχουν διαφορές. 25% στις ίδιες πολιτικές και 50% ε, για το πλάνο, για το σχέδιο Juncker. Εδώ αντιφάσκουν τα νούμερα. Επίσης θα ήθελα να πω τα εξή τα προγράμματα τα οποία πράγματα έχουν μια υπεραξία για, τον, ε, για τους πολίτες. Αναφερθήκατε σε αυτά τα προγράμματα, αλλά καμιά φορά εδώ υπάρχει μια αντίθεση. Καμιά φορά οι κλιματικοί στόχοι, ε, εάν τις ερμηνεύσουμε μη, όχι τόσο ευέλικτα, τελικά μειώνουν τις επενδύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άλλη για το Άλντε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Χόιερ, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεσή του. Ο ρόλος της τράπεζας είναι να υποστηρίζει επενδύσεις στρατηγικής σημασίας και να συμβάλλει στην ανάπτυξη, της δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη το 2015 και το 2016 ε, έκανε επενδύσεις ε, το 2,3% του ΑΕΠ και δημιούργησε πολλές θέσεις απασχόλησης. Ε, υπήρξε επιτυχής λοιπόν εκπλήρωση των πολιτικών της ΕΤΕΠ η δανειοδότηση είναι περίπου 70 δις, εκ του οποίου 90% ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ενισχυθούν στρατηγικές περιοχές, δημιουργία υποδομών, περιβαλλοντικά προγράμματα, καθώς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, πήραν οι μικρομεσαίες περίπου 40% του συνόλου, γιατί θεωρούνται ακριβώς η ρεχακαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Τα αποτελέσματα θα ήταν καλύτερα εφόσον ε, υπήρχε μια ε, εάν υπήρχε μία αύξηση συγγνώμη, της ε, χρηματοδότησης. Το Διευθυντικό Συμβούλιο της Τράπεζας ε, παρουσίασε μία έκθεση των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, στην εταιρική διακυβέρνηση θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στους μεσοπρόθεσμους στόχους όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τους σκοπούς της τράπεζας προκειμένου να αποβοηθούν ορισμένοι κλάδοι και περιφέρειες ε, που εμπίπτουν των στόχων στρατηγικής επενδύσεων. Το ΕΦΣΙ ε, βρίσκεται πολύ κοντά στην εκπλήρωση των στόχων του ε, και υπάρχει εδώ μια βελτίωση των ανισορροπιών μέσω των αποφάσεων που έλαβε το Διευθυντικό Συμβούλιο του, του ΕΦΣΙ. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Στάραντ, Σας παρακαλώ να περιοριστείτε στο χρονομιλία σας. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν ε, θα αξιολογήσω τη σύγκριση που έκανε ο, ο Δούκας του Ντάρτμουθ σχετικ... ανάμεσα στην ε, ΕΤΕΠ και την Deutsche Bank, αλλά θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που δεν συγκρίνουμε την ΕΤΕΠ με την Danske Bank, που φαίνεται ε, να έχει πολύ πιο σκοτεινό προφίλ. Παρά την άρνησή σας, κύριε Χόγερ, θα θέλαμε πολύ να δούμε τι έχει πει ο Όλαφ σχετικά με τη σχέση της τράπεζάς σας με το Volkswagen Gate. Ε, το σκάνδαλο της Volkswagen. Η διαφάνεια δεν ε, θα βλάψει ούτε εσάς ούτε εμάς. Επίσης, Οι αποεπενδύσεις φαίνονται να υπόσχονται πολλά, ε, για παράδειγμα την ε, βιομηχανία του άνθρακα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να μην επενδύουμε σε μη, βιώσιμες, σε μη βιώσιμους τομείς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τάραντ. Από την ΚΟΕ, ο κύριος Φλάναγκαν. Δύο λεπτά παρακαλώ. Με κάποιε επιφυλάξει μπορώ να στηρίξω την ε, πρότασή Σα ε, Πολύ καλή η δουλειά σα, ε, κύριε Πυρίνσκι. Η ΕΤΕΠ αποτελεί ιστορία επιτυχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα τελευταία χρόνια χαιρόμαστε που βλέπουμε να επενδύει σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων έναν τομέα που έχει εγκαταλείψει ο σημαντικό τραπεζικό τομέα όχι μόνο στη χώρα μου αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλώ με ψηφοφόρου γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει στην Ιρλανδία να βάλουν χρηματοδότηση ακόμη και για τις πιο βιώσιμες επιχειρήσεις. Οι τράπεζες έχουν ε, εγκαταλείψει την ευθύνη τους στον τομέα αυτών όπου θα πρέπει να, δίνουν, να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία. Βέβαια δεν θα χρειαζόμασταν την χρηματοδότηση αυτή υπό άλλες συνθήκες. Στην σελίδα 96 της έκθεσης για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει ότι η μείωση ε, κάποιων αξιογράφων από την Τράπεζα της Ιρλανδίας αποτελεί σημαντικό βήμα ε, για την πλήρη διάθεση των ε, στοιχείων αυτών του ενεργητικού και η υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες σχετικά με τη χρηματοδότηση. Σας μεταφράζω τα λόγια, λέει ο μιλητής. Περισσότερες επιτυχίες ε, υπάρχουν ε, το 2017. Ε, η τράπεζα της Ιρλανδίας κατέστρεψε 4 δισεκατομμύρια Είχαμε διάσωση μιας τράπεζας που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην ε, Ιρλανδική κυβέρνηση εκβιάζοντάς την. Ε, έτσι έχουν ε, ήδη χαθεί 19 δισεκατομμύρια και με σχέδια να εξαφανιστούν και άλλα χωρίς διαμαρτυρία από την Ιρλανδική κυβέρνηση. Θα ήθελα να συγχαρώ και πάλι τον κύριο Πυρίνσκι για την έκθεσή του και να ε, συγχαρώ και την ΕΤΕΠ για τη δουλειά της. Ε, θα παρακαλούσα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να λάβει γνώση αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Φλάναγκαν. Ο κύριος Άνεμανς, ένα λεπτό. Συνάδελφοι, η ΕΤΕΠ δεν θα έπρεπε να είναι ε, εργαλείο ε, της μόδας. Ε, θέλουμε εδώ να διευρύνουμε τις επενδύσεις τις πράσινες παρότι έχουν ήδη φτάσει το όριο που έχουν θέσει ήδη του 25%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κατάφερε να πετύχει ούτε τον ταπεινό στόχο του 20%. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα επενδύσει περισσότερο σε τομείς όπου υπάρχει διαφυγή εγκεφάλων φτωχές υποδομές και έλλειψη αξιόπιστων θεσμών. Αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος ε, της ΕΤΕΠ. Ε, είναι πιο πολύ να επενδύσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υποδομές κλπ. Θα πρέπει να συνεχίσει να είναι τράπεζα και να επενδύει ε, επιχειρησιακά σχέδια αντί να είναι ένα πολιτικό όχημα και γι' αυτό θα πόσχω κατά την ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ κύριε Άνεμαν. Το λόγο έχει η κυρία Γκρέσλε από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Χόιερ, Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Χαιρόμαστε που είστε εδώ και θέλω να προσπαθήσω επίσης να είμαι εντό του θέματος. Ε, πράγματι, σημειώσατε σημαντικές πρόοδους στη διακυβέρνηση της τράπεζας, γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες. Παρ' όλα αυτά, έχουμε κάποιες προτάσεις σε σχέση με τα τυχόν ε, λύματα ε, την αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας όσον αφορά τις σε τεπ, απέναντί μας κυρίως και θα ήθελα να προσπαθήσω στο χρονικό περιθώριο των διαβουλεύσεων να συμμετάσχω και εγώ. Όσον αφορά το, την αύξηση της διαφάνειας, σε επιχειρησιακό επίπεδο και τα όργανα της ΕΤΕΠ, εδώ θα πρέπει να, γίνει ε, μια, ε, να υπάρξει μια βελτίωση. Ε, και μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε για το, ε, τα διοικητικά κόστη ε, και επίσης ε, θα έπρεπε να υπάρχει μια παρακολούθηση των ε, προγραμμάτων που χρηματοδοτεί η ΕΤΕΠ καθώς και τα στοιχεία για τα ιδιωτικά κονδύλια στα προγράμματα αυτό γιατί ε, ε, έχουμε την εντύπωση ότι συχνά πρόκειται μόνο για δημόσιους πόρους. Όλα αυτά τα στοιχεία θα ήταν πολύ χρήσιμο να τα είχαμε και επίσης θα μπορούσε να είναι και μια γυναίκα ανάμεσά σας στο διευθυντικό όργανο. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκρέσλε. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Λιμπεράτσκι για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψατε μου να μην θες το ερώτημα για την ποσότητα των γυναικών. Α το αφήσουμε όσον αφορά τι τραπεζικέ υποθέσει. Είχαμε ένα καλό εισηγητή, τον κύριο Πυρίσκη, και καταλήγω στο εξή συμπέρασμα. Ένα υγιές, ένα υγιής οργανισμός, ο οποίος είναι προσανατολισμένος προς μια υψηλή επίδοση και εκπλήρωση των στόχων της. Ε, ε, και ε, η χρηματοδοτική δραστηριότητα της τράπεζας, ε, γιατί είσαστε μια τράπεζα χρηματοδότηση επενδύσεων. Και θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου όσον αφορά την ε, ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση, συγγνώμη, της ανάπτυξης. Ε, ίσως θα έπρεπε να υπάρξει και ένα συνδυασμό των κονδυλίων του ΕΦΣΥ, των κονδυλίων της ΕΤΕΚ και του ιδιωτικού τομέα, χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να αυξήσει ο χρηματοδοτικός όγκος. Το 2017 ε, το η περιφερειακή ισορροπία έχει βελτιωθεί. Αυτό θα ήθελα να κάνω μια έκκληση, όχι μόνο όσον αφορά την ε, διαβούλευση, αλλά όσον αφορά τη διεύρυνση των γνώσεων για τα σύγχρονα εργαλεία σε εκείνες τις χώρες που δεν είναι τόσο ενήμερες για αυτές τις εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λιμπεράτσκι. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Μαριάς. Για ένα λεπτό, παρακαλώ. Κύριε Χόγερ, η παροιμία λέει ότι η σιωπή είναι χρυσός. Δεν μου απαντήσατε τίποτε για τη fraport που σας είπα προηγουμένως. Ξέρετε, οι ξένοι επενδυτές πρέπει να φέρουν ζεστό χρήμα για να είναι επενδυτές. Να μην χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να κάνουν δίθεν επενδύσεις και μάλιστα να αρπάξουν δημόσια περιουσία. Δεύτερη περίπτωση. Διεθνής αερολιμένας Αθηνών. Οι διεθνεί επενδυτέ πήραν από εσά 250 εκατομμύρια ευρώ, από την ΕΤΕΠ δηλαδή, για να μπορέσουν να βρουν τα λεφτά να επεκταθεί η σύμβαση για 20 χρόνια. Ο ΤΑΠ, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ δώσατε στις πολυεθνικές στην bp και επειδή ο κύριος κατάινεν δεν κατάφερε να σας προστατεύσει διότι αυτά που δώσατε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ελληνικές είναι ψίχουλα αλλά το εύση στο οποίο λειτουργεί και η Ελλάδα και είναι πρωταθλητής ξέρετε γιατί 280 εκατομμύρια στη Fraport 150 εκατομμύρια στην Κοσμοτέ δηλαδή στην Deutsche Bank 350 εκατομμύρια σε γαλλική πολυεθνική που αγόρασε την ΔΕΣΦΑ, την εταιρεία φυσικού αερίου. 700 εκατομμύρια ευρώ του ΕΦΣΙ για τον ΤΑΠ. Γι' αυτό είναι πρωταθλητρία η Ελλάδα. Γιατί ήρθαν τα χρήματα και πήγαν στις πολυεθνικές. Έτσι είναι η κατάσταση. Να λέμε την αλήθεια. Σας ευχαριστούμε κύριε Μαριά. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Φανίστελ Ρόι. Κυρία Πρόεδρε. Κύριε Χόγερ, κύριε Επίτροπε. Κάποιες παρατηρήσεις από την προοπτική της ε, περιφερειακής ανάπτυξης. Ο κύριος Χόγερ ήδη ανέλησε τον τρόπο που εργάζεται για να ε, αποκαταστήσει την ισορροπία στην Ευρώπη, κάτι που κάνετε τα τελευταία δέκα χρόνια από, την, ε, από το ξέσπασμα της κρίσης ε, και συνεχίζετε και το κάνετε αυτό και χαίρομαι πολύ που στην έκθεση αυτή ο κύριος Πυρίνσκι έχει εξετάσει αναλυτικά την εδαφική πτυχή που είναι τόσο σημαντική στην Ευρώπη. Δεύτερη παρατήρηση, ε, ο συμβουλευτικός σας ρόλος. Ε, χθες ε, μας μιλήσατε για το EU που είναι ένας νέος κόμβος στον οποίο θα συμμετέχετε κι εσείς. Θα πρέπει να έχουμε πολύ πιο στοχευμένες εργασίες στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να έχουμε ένα καλό πρόγραμμα για τις περιφέρειες και αυτή τη στιγμή χρηματοδοτείται το πρόγραμμα, υπάρχουν σύμβουλοι αλλά δεν έχει ακόμη απογειωθεί το πρόγραμμα όπως θα θέλαμε. Φαίνεται να υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Ελπίζω ότι το InvestEU επίσης θα συμβάλλει στην πραγματοποίηση του προγράμματος αυτού. Και τρίτη παρατήρηση, έχετε κάπως λιγότερο αποκλειστική θέση ε, στο InvestEU. Ελπίζω να μπορέσετε να εργαστείτε και με άλλους εταίρους. Το InvestEU θα πρέπει να κινείται από την πολιτική. Το συζήτησαμε αυτό χθε. Θα πρέπει να λογοδοτείτε και να λογοδοτείτε και για άλλα προγράμματα. Αλλάζει ο ρόλος σας και η κυρία Γκρέσλε έχει δίκιο. Θα πρέπει να ασχοληθείτε και με την διακυβέρνηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Φανίστελ Ρόι. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Κέλλη, παρακαλώ. 1,5 λεπτό. Δεν σας βλέπουμε πολύ, πολύ συχνά. Γιατί δεν είναι εδώ ο χώρος, το χώρος εργασίας σας. Γι' αυτό είναι ευχάριστο που είστε σήμερα εδώ, κύριε Χόγη, και μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψει μαζί σα, ε, αλλά και να σα χαρούμε για την καλή δουλειά που έχει κάνει η ΕΤΕΠ προωθώντα τι επενδύσει και που οδηγού, πράγμα που οδηγεί στην ανάπτυξη και την ευημερία. Σε 60 χρόνια έχετε επενδύσει σε 160 χώρε και είναι εντυπωσιακό ε, το ε, ρεκόρ σας. Ιδιαίτερα ο ρόλος που παίξατε τα τελευταία χρόνια της ύφεσης είναι πολύ σημαντικός και νομίζω πως ανοίξατε και ένα γραφείο στο Δουβλίνο με τον κύριο Κόνον Μέρφυ επικεφαλής και θέλω και εκείνον τον συγχαρώ για την καλή τη δουλειά και για τη συνεργασία με μένα αλλά και τον Επίτροπο Κατάινεν που διοργάνωσε διάφορα σεμινάρια στο υπεριφέρειά μου για το ΕΦΣΥ με μεγάλη επιτυχία όπως ε, τονίσατε και εσείς και είμαι ευτυχής πως εισηγητής για την Επιτροπή Βιομηχανίας μπορώ να σας πω πως ε, ε, ε, <clears throat> υπερψηφίσαμε τη συνέχιση του InvestEU. Θέλουμε να ε, τονιστεί περισσότερο η στήριξη των μικρομεσαίων. Εν γέννη λοιπόν γίνεται πολύ καλή δουλειά. Καλωσορίζω τα όσα είπατε για το Brexit, αλλά ελπίζω πως τα κράτη-μέλη θα δείξουν την ίδια γενοδορία στο να καλύψουν το κενό που θα αφήσει το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με το γενικό μας προπολογισμό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Και τώρα θα περάσουμε στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Στρογεύσκη είναι ο πρώτος ομιλητής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, τέσσερα σημαντικά σημεία το ΕΦΣΙ έχει μια καλή ε, ε, ε, δράση. Και γι' αυτό χαιρόμαστε. Ωστόσο, η διαδικασία της μόχλευσης δεν είναι έτσι όπως την είχαμε προβλέψει. Ίσως υπήρξαμε υπερβολικά αισιόδοξοι. Οι γεωγραφικές ανισορροπίες έχουν αποδυναμωθεί μεν, αλλά όλη αυτή η διαδικασία είναι αρκετά βραδία Επίσης, όσον αφορά τις επενδύσεις στις διατησιμικές τεχνολογίες, εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Τα όσα ακούσαμε μέχρι στιγμής ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Ο κύριος Πρόεδρος Ε, υπερεύει το χρόνο του, ενώ ο κύριος Κατάινεν χρησιμοποιήσει μόνο το 60% του χρόνου του. Αλλά χρειαζόμαστε περισσότερες ε, διευκρινήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πόλτσακ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζω την κατάσταση της ΕΤΕΠ καθήκον της είναι να επενδύει στρατηγικά ε, σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Θα ήθελα να συμφωνήσω και με την αξία της ε, γεωγραφικής ισορροπίας και γεωγραφικής συνοχής θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όσον αφορά την ετήσια έκθεση, το 40% των επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είχαν στόχο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε νομίζω ότι έχει πετύχει τον σχετικό της στόχο η τράπεζα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τη δανειοδότηση. Πρέπει να γίνεται αποτελεσματικά, αλλά με την αστάθεια που επικρατεί στις αγορές ε, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, κάτι που δεν έχουμε δει εδώ ακόμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πόλσακ. Δίνω το λόγο στον Επίτροπο Κατάινεν. Παρακαλώ. Θα ήθελα να επενέσω την δουλειά του ε, κυρίου Κέλλη στην εκλογική του περιφέρεια. Ξέρω ότι δεν είναι ο μόνος, αλλά θα ήθελα ε, να αναφέρω τη δουλειά που έχει κάνει ως υπόδειγμα. Κάτι τέτοιο ακριβώς χρειαζόμαστε. Χρειάζεται να πούμε στους πολίτες μας και στις επιχειρήσεις μας τι υπάρχει, τι ε, διατίθεται, πώς μπορούν να υποφεληθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τι έχει να τους προσφέρει, διότι αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να μην γνωρίζουν οι πολίτες τι υπάρχει, τι δυνατότητες υπάρχουν. Δεν είναι πολύ εύκολο να καταλάβει κανείς ε, τα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων όσο είναι να καταλάβει τα δάνεια μιας ε, σημαντικής τράπεζας. Ε, πρέπει να ενημερώσουμε τους ανθρώπους και η άνηση γεωγραφική κατανομή οφείλεται ενδεχομένως στην, στην ανισορροπία στην ενημέρωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ευρωβουλευτές για την ε, πολιτισμένη και ουσιαστική συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό. Αποτελεί πολύ καλή βάση για τη συνέχιση της συνεργασίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Χόγερ έχει το λόγο, πρόεδρος της ΕΤΕΠ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω ένα δίλημα. Μόλις με επέκριναν επειδή ε, έχω μιλήσει παραπάνω από το χρόνο που μου δώσατε, αλλά έχω 20 ερωτήσεις και πρέπει να απαντήσω. Οπότε, ε, συγχωρήστε με, αλλά θα σας απαντήσω καταλήλως όσο γίνεται πιο σύντομο. Το θέμα της περιφερειακής κατανομής αρχίζει να με εκνευρίζει, διότι πιστεύω ότι όλοι όσοι έχουν την αίσθηση ότι η χώρα τους έχει πάρει λιγότερα ή περισσότερα από τον γείτονα, μιλάει για περιφερειακή κατανομή. Σας είπα τα στοιχεία για τα project του ΕΦΣΥ. Εν γέννη, για όλα τα προγράμματα της ΕΤΕΠ βασιζόμαστε στο, GD, στο ΑΕΠ. Η Ελλάδα είναι η πρώτη, δύο είναι η Κύπρος, τρία είναι η Πορτογαλία, τέσσερα η Κροατία, πέντε η Πολωνία. Μα είναι τόσο λάθο αυτό. Αυτέ είναι οι προτεραιότητε που περιμένετε από εμά και νομίζω πως κάνουμε σημαντική πρόοδο σε αυτό το θέμα. Δεύτερο, θέλω να, να, δώσω, να, βάλω στη συζήτηση τη λέξη υποδομές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προβλήματα με την ποιότητα των υποδομών. Δεν επενδύουμε αρκετά στη συντήρηση των υποδομών μας, πράγμα που οδηγεί σε διαφορετική υποβάθμιση της ποιότητας των υποδομών μας και πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε. Πολύ πιο ωραίο είναι να χτίζουμε νέα πράγματα από ότι να συντηρούμε τα παλιά. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε για τις startups. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα για την ε, χρηματοδότηση επιχειρήσεων στην Ευρώπη και κυρίως για την χρηματοδότηση των startup. Ε, ε, αυτό γίνεται μέσα από τις τράπεζες και όχι από τις κεφαλαγορές, ενώ στη ΣΥΠΑ είναι τελείως ανάποδο. Γι' αυτό και κάποιες φορές κάποιους εφηείς εφευρέτης Μόλις αναπτύξει κάτι, ανοίγει την, μια αναγορά, αναπτύσσει ένα νέο προϊόν και αυτό ή αυτή μπορεί να έχει μεγάλη επιτυχία στην αρχική φάση και μετά έχουμε το αναπτυξιακή χρηματοδότηση και δεν έχουμε ένα τέτοιο μέσο. Πολύ θα μου άρεσε να αναπτυχθούν περισσότερο οι δραστηριότητε τη ΕΤΕΠ σε αυτό το τομέα, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου που πολλέ φορέ τα πολλά υποσχόμενα προϊόντα αναπτύσσονται εκτό ε, τη Ευρωπαϊκή Υπήρου με πολλά χρήματα. Ε, και έπειτα μετρώμε όσο γίνεται περισσότερο τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας. Να σας δώσω κάποια νούμερα αργότερα. Αλλά για παράδειγμα, στην ανάλυση μας βλέπουμε ότι το 2018 ο αριθμός των μικρομεσαίων που στηρίχτηκαν ήταν, ε, ε, ήταν 200.000 και ίσως θα έπρεπε να δίνουμε μεγαλύτερη δημοσιότητα σε αυτά μας τα νούμερα. Χρηματοδότηση, μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Κυρίε και κύριοι, ορισμένοι θέλετε να μας δείτε ως εμπορική τράπεζα και άλλοι ως πολιτικό μέσο. Είμαστε και τα δύο. Πρέπει να λειτουργούμε σε διάφορους τομείς ως σαν εμπορική τράπεζα γιατί επαναχρηματοδοτούμε τελείως τις κεφαλαιορές. Πρέπει να έχουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών γιατί διαφορετικά δεν θα μας δώσουν 60, 70, 80 δις ετησίως. Δεύτερον, εξυπηρετούμε έναν δημόσιο στόχο. Οι στόχοι μας ορίζονται από εσά και το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνδυάσουμε το ρόλο ενός δημόσιου θεσμού με εμπορική συμπεριφορά και εμπειρογνωμοσύνη στις αγορές. Και νομίζω πως το καταφέρνουμε αρκετά καλά. Για το θέμα της διαφάνειας, κυρία Γκρέσλε, Συμμερίζομαι τη γνώμη σας και νομίζω πως προοδεύουμε, αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε και καλύτερα. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα, μάλλον δύο, που θέλω να πω. Ε, πρώτον, να έχετε υπόψη ότι η ΕΤΕΠ είναι πολύ ε, ε, σπαρτιάτικο ίδρυμα. Έχουμε 3.000 υπαλλήλους. Ακούγεται πολύ, αλλά δεν είναι ε, γιατί ο όγκος, ε, η Παγκόσμια Τράπεζα έχει 18.000 ε, κόσμο. Δεν είμαστε και τόσο σπάταλο. Κάποιες φορές μας επικρίνουν ότι δεν εκπροσωπούμαστε σε όλες τις χώρες της Ένωσης με επίσημα γραφεία. Προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί. Παρακαλώ αυτό να το θεωρήσετε ως μια σοβαρή προσπάθεια να είμαστε ορατοί και διαθέσιμοι παντού, αλλά το κόστος, ε, η μείωση του κόστους ή, εν περιπτώσει, ο περιορισμός του κόστους είναι μια στρατηγική που την ε, ακολουθούμε. Και τέλος για το φίλο, κυρία Γκρέσλε. Κοιτάξτε, χτυπάτε ανοιχτέ πόρτε. Οποτεδήποτε έρχεται ένα κράτο μέλο με νέα πρόταση για το διοικητικό ε, και η Επιτροπή και κάποιο κράτο μέλο προτείνει μια κυρία με μεγάλη χαρά θα την υποδεχτούμε. Η Ισπανία μόλις το έκανε και σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες γυναίκες. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται από εμά, εξαρτάται αποκλειστικά από τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά το επικεφαλής μας διοικητικό προσωπικό, τα τελευταία χρόνια από 18% έχουμε φτάσει στο 26% στις ε, ανώτατες θέσεις. Προχωράμε. Δεν μπορεί αυτό να γίνει σε μία νυχτή γιατί χρειάζεται ένα-δύο χρόνια στα διαδρομία στην τράπεζα για να φτάσει κανείς σε top θέσεις. Αλλά το έχουμε υπόψη μας. και το επιδιώκουμε, χωρίς βέβαια να επιβαρύνουμε το άλλο φύλλο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενικέ ε, Διοικητή. Θα σας τονίσω ότι δεν είμαι βέβαιος ότι ο βέβαια ότι ο κύριος Στρογεύσκη ήθελε να μιλήσετε λιγότερο. Ίσως θέλατε... ήθελε να μιλήσει περισσότερο ο αντιπρόεδρος Κατάινεν. Μεγάλο μας τιμή που είστε σήμερα εδώ. Και τώρα θα καλέσω τον εισηγητή μας, κύριο Πυρίσκη, να κλείσει την συζήτηση ε, παίρνοντας και εκείνο το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους σχολιάσαν την έκθεση. Θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι μια έκθεση του συνόλου της Επιτροπής και ε, τα όσα είπε ο κύριος Χόιερ, δηλαδή ότι τα βήματα προς την κατεύθυνση της άξιση λογοδοσίας και μεγαλύτερης διαφάνειας είναι υπόδειγμα, ε, απόδειξη χρησιμότητας ε, συζητήσεων σαν αυτές που γίνονται στην Επιτροπή μας. Επίσης θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της γεωγραφικής διάστασης αναφέρθηκαν αριθμοί που δείχνουν που δίνουν ένα μας σε ανησυχίες. Ωστόσο, μια αναλογία 80 προς 10 είναι τίποτα άλλο παρά μια βιώσιμη ισορροπία και σίγουρα μια πρόκληση στην οποία θα πρέπει να ανταπεξέλθουμε. Και τέλος θα ήθελα να αναφέρω ότι το είδος συζήτηση που κάναμε, το γεγονός ότι ο πρόεδρος ε, ήταν όσο πιο ανοιχτός ε, μπορούσε. Νομίζω ότι είναι θετικό, ναι, ε, θετικό, θετική ένδειξη όσον αφορά την πρόοδο που έχει γίνει. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Πυρίνσκι. Και εδώ κλείνει η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Και τώρα θα ήθελα να πω το εξή. Μετά τις διαβολεύσεις με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος θέλει να υποβάλει την εξή πρόταση αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Ε, την Πέμπτη ε, να γίνει ε, μία αναβολή. No, don't seem so. So τη, συζήτηση για το Τόγκο. Έχετε εδώ αντιρρήσεις. Όχι. Ωραία λοιπόν. Τώρα θα συνεχίσουμε με την ημερήσια μας ε, διάταξη. Επόμενη έκθεση είναι η έκθεση της κυρίας Καρθία Θαμπάλ Ρουμπιάλ και του κυρίου Σαρβαμά όσον αφορά ε, για την προστασία του προπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση γενικευμένων ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου στα κράτη-μέλη. Ε, καταρχήν, η οι συγητές έχουν το λόγο, η κυρία Γκάρθια Μπάλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κάποιος ε, ε, θα ήθελα να πω τα εξή. Ε, έχουμε συζητήσει πολλέ, κατ' επανάληψη τα ζητήματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπουμε πόσο αναποτελεσματικά είναι τα όργανα τη Θεσμική Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε κάποιε κοινέ αξίε που θα πρέπει να σεβόμαστε ω πολίτε και ω χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή δεν είναι μια Ευρώπη αλλά καρτ όπου μπορούμε όπου έχουμε τη δυνατότητα να μην εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας και να έχουμε μόνο δικαιώματα. Έχουμε υποχρεώσεις ε, πολιτικές, δημοσιονομικές ε, κλπ. Ε, αυτή τη στιγμή ε, έχουμε εγκρίνει τον προπολογισμό, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όχι, η εξέταση, ο έλεγχος πρέπει να είναι συνεχής. Και θα πρέπει να δημιουργηθεί και ένα σύστημα επιβολής ε, κυρώσεων. Ωστόσο, η συνθήκη δεν το προβλέπει. Γι' αυτό θα ήθελα, γι αυτό θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή έκανε μια έξυπνη πρόταση, ε, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που έχει ε, στη διάθεσή, διάθεσή της, τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Ωστόσο, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχασε μια ευκαιρία γιατί εάν συνδυάσουμε αυτέ τι δύο ιδέε, δηλαδή το σεβασμό των αξιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την προστασία του προπολογισμού, ε, δεν επαρκεί να αναφερθούμε μόνο στο κράτος δικαίου, γιατί τα, οι αξίες αυτές αναφέρονται στο άρθρο 2 της Ευρωπαϊκής ε, Συνθήκης όσον αφορά τη σεβασμό της ανθρώπινης εξωπρέπειας, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα, ελεγγύη, δικαιοσύνη, ενοχή κλπ. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 2 και ορίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι αυτά τα οποία οι αξίες πρέπει να προστατεύσουμε. Σωστά θα πρέπει να προστατεύσουμε επίση και τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη επίθεση στους, ε, στα δημόσια οικονομικά, στην αλληλεγγύη και τις ευρωπαϊκές αξίες από την ε, απάτη και την ε, φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει οι αξίες αυτές και τα κριτήρια να ελέγχονται. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ισότητα, δικαιοσύνη, ελεγγύη εάν κλείνουμε τα μάτια όσον αφορά την δημοσιονομική δικαιοσύνη. Και όπως γνωρίζετε πριν γίνει η συζήτηση για τον ε, κανονισμό, διαπραγματευτήκαμε τρία, τρεις πτυχές την ε, προστασία των τελικών παραληπτών. Ε, κάποιε κάποιες ε, κυρώσεις θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με του μηχανισμού και να εξασφαλίζουμε οι κυρώσει αυτέ ε, να επιβαρύνουν αυτού που έκαναν τι παραβιάσει και όχι του τελικού παραλήπτε. Και πιστεύω ότι χάρη στι τεχνικέ υπηρεσίε της Επιτροπής μπορέσαμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Το δίκτυο ασφαλείας που έχουμε ορίσει αποτελεί μια εγγύηση για του τελικού παραλήπτε. Το δεύτερο στοιχείο είναι το πάνελ των εμπειρογνώμων γιατί η λήψη των αποφάσεων θα είναι ένα θέμα, είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει στη διάθεσή της όλες τις ε, αναγκαίες πληροφορίες για να μπορεί να πάρει μια απόφαση αντικειμενική, ε, δικαιολογημένη και δικαιολογημένη. Και αυτό είναι ο στόχο σύσταση του πάνελ των εμπειρογνωμόνων που μπορούν να συντρέξουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τρίτον, ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, δεν θα πρέπει να περιορίσει στο ρόλο του παρατηρητού γιατί μιλάμε για αξίες στον προπολογισμό. Και όσον αφορά τον προπολογισμό, το σώμα αυτό είναι αρχή αρμόδια επί του προπολογισμού, όπω είναι και το Συμβούλιο. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγω, μια φράση που ανέφερε ο Πέδρο Σάντσεθ ε, σήμερα. Έχει έρθει η στιγμή να υπερασπίσουμε τις ε, αξίες που καθιστούν το εγχείρημά μας μοναδικό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρδιά Σαβάλ. Σάρβαμα, τέσσερα λεπτά, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η δημοκρατία ποτέ δεν είναι αυτονόητη. Ποτέ. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, αν όχι το πιο σημαντικό για τη διατήρηση της δημοκρατίας σε οποιοδήποτε κράτος, είναι ε, το κράτος δικαίου. Εάν αμφισβητείτε το κράτος δικαίου, είναι πια ανοιχτός ο δρόμος ε, για το κουτί της Πανδώρας, διότι, συνάδελφοι, η δημοκρατία ποτέ δεν είναι τέλεια. Η δημοκρατία με τις εκλογές ε, μπορεί ε, να οδηγήσει στην εκλογή ε, κυβερνήσεων και ηγετών που θέλουν να αρπάξουν το κουτί της Πανδώρας για να δουν αν μπορούν να το ελέγξουν καθοδόν ε, μπορεί να παρέμβουν ε, στους μηχανισμούς ε, του κράτους δικαίου ή μπορούν να φροντίσουν οι δημοσιογράφοι να μην θέλουν να κατακρίνουν τους, έχοντες, τους κατέχοντες στην εξουσία. Με όλους αυτούς τους τρόπους οι κυβερνήσεις και οι ηγέτες τους υπονομεύουν το κράτος δικαίου που είναι ο κεντρικός πυλώνας της δημοκρατίας. Αυτό δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι, αποτελεί περιγραφή αυτού που γίνεται σήμερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν λοιπόν θέλουμε να προστατεύσουμε τη δημοκρατία αυτή καθ' αυτή, θα πρέπει να προστατεύσουμε το κράτος δικαίου. εδώ και χρόνια είναι σαφές, επώδυνα σαφές, ότι ε, οι ισχύοντες μηχανισμοί εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ε, σταματούν ε, τις κυβερνήσεις, δεν εμποδίζουν τις κυβερνήσεις από το να ακολουθήσουν αυτόν τον επικίνδυνο δρόμο. Και γι' αυτό έχουμε μπροστά μας αυτόν τον πολύ σημαντικό κανονισμό. Χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό που θα εισάγει συγκεκριμένες συνέπειες για τα κράτη-μέλη αυτά. Και γι' αυτό πολύ σοφά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολούθησε την επιθυμία του Κοινοβουλίου ε, το ψήφισμα ε, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο του Κοινοβουλίου ε, και εισάγει έναν μηχανισμό για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης στην περίπτωση ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να επιβάλλει κατάλληλα μέτρα για τον ε, περιορισμό ή την ε, αναστολή της πρόσβασης σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με τρόπο ανάλογο με την ε, φύση και την σοβαρότητα και το εύρος των ελλείψεων. Πέντε πράγματα θα ήθελα να τονίσω για να καταλάβετε αυτή την νομοθετική έκθεση. Η νομική βάση της πρότασης αυτής είναι ο δημοσιονομικός κανονισμός και όχι το άρθρο 7. Ε, μιλάμε για προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης, δηλαδή των ε, χρημάτων ε, των φορολογουμένων. Δεύτερον, θέλουμε να συντάξουμε ένα νόμο που να ισχύει ίσα για όλα τα κράτη-μέλη. Μπορεί να έχουμε παραβίαση του κράτου δικαίου σε οποιοδήποτε κράτο μέλο. Τρίτον, θέλουμε να προστατεύσουμε τους τελικούς δικαιούχους ε, της Ευρωπαϊκής ερευνητέ, ερευνητές, οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών. Οι κανονικοί πολίτε δεν θα πρέπει να υποφέρουν από τον περιορισμό τη χρηματοδότηση. Τέταρτον, μιλάμε για γενικευμένε ελλείψει όσον αφορά το κράτο δικαίου. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουμε σαφή και ευρία υπονόμευση του κράτου δικαίου προτού να μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία κυρώσεων. Και πέμπτον, το Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο θα λαμβάνει αποφάσεις σε ε, ίση βάση. Με τα λόγια μου αυτά, ελπίζω κάθε μέλος του Κοινοβουλίου να ε, εξετάσει προσεκτικά την έκθεση αυτή. Και πιστεύω ότι θα ε, θεωρήσετε σημαντικό να στηρίξετε την πρόταση αυτή και να μας δώσετε ισχυρή εντολή για τον τριμερή διάλογο, διότι Τίποτα, τίποτα ε, στη σημερινή Ευρώπη δεν είναι τόσο σημαντικό όσο είναι το κράτος δικαίου. Και τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, και να επενέσω την ε, συνεισηγήτριά μου, την κυρία Γκουαρδία Σαβάλη, για την εξαιρετική εργασία που έχει κάνει στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σάρβαμα. Από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, η κυρία Σαρτζεντίνη, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ αντικαθιστώ τον κύριο Τέρι Κάμπρα, τον συνάδελφο που είναι αρμόδιος για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας. Είμαι και εγώ επιβεβαισμένη ότι αυτή η πρόταση είναι απαραίτητη. Οφείλουμε να φτιάξουμε όλα τα απαραίτητα <clears throat> μέσα για να εγγυηθούμε το σεβασμό του νόμου στα κράτη-μέλη. Είναι ρόλος μας να προστατεύσουμε του Ευρωπαίου πολίτε σε σχέση με, απέναντι στι κυβερνήσει που μπορεί να καταπατούν τα ατομικά δικαιώματα. Θα πρέπει ε, Όντω, οι ευρωπαϊκέ επιδοτήσει να εξαρτώνται από το σεβασμό του κράτου δικαίου. Αυτό το νέο μέσο ήταν απαραίτητο για να εγγυηθούμε το σεβασμό του δικαίου. βλέπω και σκέφτομαι κυρίως στην Ουγγαρία, βλέπω και κυβερνήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση που προσπαθούν να, να, να το καταπολεμήσουν αυτό. Δεν πρέπει να μείνουμε ε, απαθείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εγγυηθεί τα δικαιώματα των ε, πολιτών. Έχουμε το χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουμε το κράτος δικαίου. Ε, τροπολογία 72 του εισηγήτρια πιστεύω πω βελτιώνει την έκθεση και την υποστηρίζουμε. Σα ευχαριστούμε. Και σας ευχαριστούμε πολύ που μας θυμίζετε ότι πρόκειται ε, για δουλειά του κυρίου Τέρι Κάμπρας. Τον λόγο έχει ο Επίτροπος Έτινγκερ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν θα ήθελα εκ μέρους της Επιτροπής να ευχαριστήσω όλους ε, τους συγητές, ε, την κυρία Γκαρθιαμπάλ και τον κύριο Σαρβάμαν, αλλά και εσάς κυρία Σαρκεντίνη, για την ε, εξαιρετικά τεκμηριωμένη ε, ανασχόληση με την πρόταση, την οποία δέχεστε κατ' ουσία, αλλά θέλετε να επιφέρετε κάποιες βελτιώσεις. Ε, η πρόταση κανονισμού της Επιτροπής αφορά τις ε, γενικευμένες ελλείψεις σε σχέση με το κράτος ε, δικαίου στα κράτη-μέλη και σε συνάρτηση βεβαίως με τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ε, θέμα είναι να δημιουργηθεί ένα εργαλείο το οποίο να εξασφαλίζει τους ε, πολίτες από φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και φοροαποφυγής και διαφυγής σε συνεργασία με το Συμβούλιο. Ένα τέτοιο εργαλείο έχει μεγάλη σημασία. Ε, θα έπρεπε ήδη να έχει συσταθεί. Το ότι το προτείνουμε είναι απολύτως εύλογο, γιατί στα προγράμματα του προπολογισμού, εκεί που θέλουμε να προωθήσουμε κάποια προγράμματα ή που εγκρίνουμε κάποιες ε, προτάσεις ή εκταμεύονται χρήματα, ε, υπάρχει το θέμα ε, των ε, παραληπτών και αντιπαραθέσεις με περιφέρειες, ε, δήμους, χώρες κλπ. Θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στις χώρες μέλη όσον αφορά την ανεξαρτησία των δικαστηρίων. θα πρέπει ε, το κράτος δικαίου λοιπόν να έχει απεριόριστη ισχύ σε όλες τις χώρες ε, μέλη. Και ήδη τώρα οι χώρες μέλη πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι διατάξεις τους για όσον αφορά την απορρόφηση των ε, οικονομικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αποτελεσματικά και υπάρχει επαρκής προστασία εναντί φαινομένων απάτης. Εμείς με την πρόταση αυτή ενισχύουμε τα εργαλεία μας και αυξάνουμε και την, ενισχύουμε την υπόλοιψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένας τέτοιο μηχανισμός για την προστασία των χρημάτων των ε, πολιτών και φορολογουμένων μας ε, σε σχέση με γενικευμένες ελλείψεις όσον αφορά το κράτος δικαίου σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Η, ο ε, η εστίαση μάλλον στην αρχή του κράτους δικαίου είναι αρθή. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει ορισμός του πεδίου εφαρμογής να γίνει προσεκτικά ε, και μάλιστα σε σχέση με άλλους μηχανισμούς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα το άρθρο 7 της συνθήκης. Γιατί δεν πρόκειται για την επιβολή κυρώσεων εδώ, αλλά πρόκειται για την προστασία των ευρωπαϊκών χρημάτων και, καθώς και για την ορθότητα της εκτέλεσης του προπολογισμού σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή προτείνουμε έναν διαφανή και αντικειμενικό μηχανισμό και τα τυχόν μέτρα θα πρέπει να είναι σε μία αναλογία με, το, με την φύση και την ε, βαρύτητα των ε, παραβιάσεων των αρχών του κράτους δικαίου, δηλαδή περικοπές ή ε, κατάργηση ή ε, ε, μη εκταμίευση των κονδυλίων σε αναλογία, όπως είπα, της βαρύτητας της παραβίασης όσον αφορά τις αρχές του κράτους δικαίου. Γιατί ο πολίτης, ο, ο, ο αποδέκτης δεν θα πρέπει να είναι ο βλάκας. Θα πρέπει οι πολίτες και τα προγράμματα να λάβουν τελικά αυτά ε, που ε, τους ανήκουν. Ε, δεν θα πρέπει δηλαδή να είναι εις βάρος της κοινωνίας, των σπουδαζόντων, των υπαλλήλων κλπ. Εάν η Επιτροπή έχει λόγους να πιστεύει ότι διαπιστώνεται έλλειμμα αρχών του κράτους ε, δικαίου ε, θα ε, κινήσει μια διαδικασία που μπορεί να οδηγεί στη λήψη των δεγμένων μέτρων. Θα πρέπει να λάβουμε εδώ υπόψη μας τις αποφάσεις του δικαστηρίου, εκθέσει του ελεγκτικού συνεδρίου, καθώς και πορίσματα αρμόδιων ε, οργαν, οργανισμών. Πριν λάβουμε την απόφαση θα πρέπει να κάνουμε μια ακρόαση, θα πρέπει να ακούσουμε μάλλον την ε, ε, ε λόγω την κατηγορούμενη χώρα. και η διαδικασία λήψης ε, απόφασης θα πρέπει να είναι ταχεία και αποτελεσματική, μη γραφειοκρατική